Good morning, dear colleagues. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Η κυρία Μανέσκου μπλέχτηκε στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα καθυστερήσει λίγο. Οπότε, εν αναμονή τη κυρία Μανέσκου, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο τη διάταξης, διάταξη, την επίτευξη της πραγματικής εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απαραίτητη προπόθεση για την ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο επίπεδο. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λούχαν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. E Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ενδεικτικό τη σημασία που προσδίδουμε στην εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή το γεγονό ότι ασχολούμαστε με την έκθεση αυτή. Εγώ στην έκθεσή μου θα αναπτύξω κυρίως αυτό που λέει ο τίτλος της έκθεσης, την επίτευξη της ουσιαστικής εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, που είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα στο παγκόσμιο επίπεδο. Θα δούμε ποιες είναι οι προοπτικές ε, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσω έμφαση στο ρόλο που διαδραματίζει για την ανταγωνιστικότητα αυτή η συνοχή. Πιστεύω ότι μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να κατευθύνουμε τις εσωτερικές μας πολιτικές προς αυτό το στόχο. Και θα πρέπει να διαρωτηθούμε πώς θα καταστήσουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική διεθνώς και πώς θα επιλύσουμε τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας πέραν της ε, σοβούσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές σημαντικές προκλήσεις. Την προσαρμογή μας στην παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές και τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και διάφορα ενεργειακά ζητήματα. Όλα αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το 2020. Και προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο όλων αυτών των προκλήσεων στους Ευρωπαίους πολίτες, θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο των περιφερειών σε αυτή την προσπάθεια και το πώς θα μπορέσουμε εμείς να στηρίξουμε στο έργο τους περιφέρειες. Για να ελοπίσουμε τους στόχους της στρατηγικής του 2020, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ξεκινάμε από διαφορετικά αναπτυξιακά επίπεδα στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Γι' αυτό και θα πρέπει να θέσουμε ρεαλιστικούς στόχους που θα στηρίζονται στην ε, πραγματικότητα της κάθε περιφέρειας και φυσικά θα προσαρμόζονται στην πολυεπίπεδη αυτή διακυβέρνηση. Η έκθεσή μου χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα. Το πρώτο τμήμα, όπως θα είδατε, αφορά κάποια γενικά θέματα για την ε, ανταγωνιστικότητα στα οικονομικά θέματα. Το δεύτερο τμήμα αφορά την εδαφική συνοχή και τον αντίκτυπο της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής στη συνοχή αυτή. Το τρίτο τμήμα μιλά για την ε, μεγιστοποίηση του αντικτύπου της πολιτικής συνοχής προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και το τελευταίο τμήμα της έκθεσής μου μιλά για την περίοδο μετά το 2013 σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Η έκθεση αυτή εκπονήθηκε χάρη σε πολλές ε, πληροφορίες και πηγές που αναφέρω στην αρχή της έκθεσης και μάλιστα οι αιτήσεις εκθέσεις του Παγκόσμιου Φόρουμ ήταν πολύ σημαντικό για θέματα παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και περιμένουμε και την, ε, το χειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα που θα ακολουθεί την γενική προσέγγιση του, της απογραφής για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Χρησιμοποίησα και την έκθεση του ΩΣΑ για την οικονομική συνεργασία και την ανάπτυξη και έλαβε υπόψη και το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη στον ΩΣΑ. Για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ανταγωνιστική και διεθνώ, θα πρέπει να ενισχυθεί πρώτα στο εσωτερικό τη. Και το θέμα είναι πώ θα καταφέρουμε κάτι τέτοιο, πώ θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Το σχέδιο εκθεσή μου υποβάλλει κάποιε προτάσει σχετικά. Καταρχήν, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε παρόμοιο βιωτικό επίπεδο σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Δηλαδή, θα πρέπει να στηρίξουμε τις περιφέρειες και να τις χρηματοδοτήσουμε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους και τις ανάγκες τους. Έτσι θα βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των τοπικών πόρων και θα αναπτύξουμε το τοπικό δυναμικό. Επίσης θα πρέπει σε περιφερειακό πάλι επίπεδο να υποστηρίξουμε την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη και την έρευνα. Και επίσης θα πρέπει να δώσουμε τους καρπούς της Ευρωπαϊκή πολιτική τη συνοχή. Γιατί αν αποτύχει η πολιτική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτύχει και ο στόχο μα τη ανταγωνιστικότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εδαφική συνοχή είναι επίσης ε, μια κοινή βάση και σημαίνει πρόσβαση όλων των πολιτών στις υποδομές και στις υπηρεσίες η εδαφική συνοχή θα είναι η, ο κραγωνιαίος της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. Και χάρη στην πολιτική συνοχής θα έχουμε μια προστιθέμενη αξία και στα θέματα της ανταγωνιστικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα ξεκίνησε και ο διαρθρωτικός διάλογος με την Κίνα αρχικά και με τη Ρωσία αργότερα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε τα ωφέλη της πολιτικής συνοχής, αλλά το θέμα είναι με ποιο τρόπο. Καταρχήν, προσπαθώντας να πλουστεύσουμε τις εφαρμοστικές διαδικασίες για τα σχέδια και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα διευθυντικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Επίσης, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητα αυτών των προγραμμάτων. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερο την αρχή της εταιρικότητας και να ενισχύσουμε το δυναμικό των θεσμικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει να κρατήσουμε το ΑΕΠ ως βασικό δείκτη για την κατανομή των διαρθρωτικών κονδυλίων και των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειές μας θα πρέπει να γίνουν και προκλήσεις της πολιτικής συνοχής. Από αυτή την άποψη η πολιτική συνοχή θα είναι κέρια πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, οι περιφέρειες τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διαφορετική δυνατότητα αντίδραση, αλλά έχουν κοινά προβλήματα. Για παράδειγμα, τι κλιματικέ αλλαγέ θα πρέπει να τι καταπολεμήσουμε με μια κοινή προσέγγιση. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε τη συνοχή. Θα πρέπει επίση να συνεχιστεί η διαδικασία αποκέντρωση στα κράτη-μέλη και να δοθούν περισσότερε εξουσίε και αρμοδιότητε περιφέρειε προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλε αυτέ τι προκλήσει. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το διοικητικό τους δυναμικό για να μπορέσουν και οι περιφέρειες να διαχειρίζονται όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των διαρθρωτικών κονδυλίων στο μέλλον. Έτσι θα αισθανθούν καλύτεροι οι πολίτες και τα πραγματικά ωφέλη της πολιτικής συνοχής, μια και αυτή θα τη διαχειρίζονται οι περιφέρειες και η τοπική αυτοδιοίκηση που είναι πολύ πιο κοντά στους πολίτες. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις διάφορες υποδομές στις μεταφορές, παιδεία, υγεία και να εξασφαλίσουμε πρόσβαση όλων των πολιτών σε υποδομές αυτές. Έτσι θα βελτιωθεί το βιωτικό τους επίπεδο και θα μεγιστοποιήσουμε και το αναπτυξιακό τους δυναμικό. Βέβαια, οι τοπικές και περιφερειακές ε, τάσεις θα εξαρτηθούν από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και της κάθε περιφέρειας. θα πρέπει να βελτιωθεί η ανάπτυξη στις περιφέρειες και να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους, γιατί δυναμικό υπάρχει και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της αλληλεγγύης και της οικονομικής ισορροπίας. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και την αλληλεγγύη και μια οικονομική ισορροπία και αυτό θα γίνει χάρη σε κοινέ προσπάθειες και σε μακροπρόθεσμες προοπτικές. Φυσικά δεν είναι τέλεια η έκθεση, επιδέχεται βελτιώσεις και βλέπετε ότι ο τίτλος προδίδει ένα ευρύτατο πεδίο, γι' αυτό έκανα στην αρχή κάποια γενικά σχόλια, αλλά μετά επικεντρώθηκε σε τρεις συγκεκριμένους τομείς για τους οποίους υπέβαλα και αυτές προτάσεις προκειμένου να φανεί προς τη θέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής. Περιμένω τα σχόλιά σας αγαπητοί συνάδελφοι, τις προτάσεις σας και τις ιδέες σας για να εμπλουτιστεί το σχέδιο εκθεσής μου. και πιστεύω ότι αυτή η έκθεση για την πολιτική συνοχή θα δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να δρέψουν και οι συμπολίτες μας τους καρπούς της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ και περιμένω τις τροπολογίες και τις προτάσεις. Okay, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η έκθεση τίθεται προς συζήτηση. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε ιδιαίτερα γιατί ξεκαθαρίστηκε το θέμα. Ο τίτλος εκπλήσει κάπως, όλα τα άλλα είναι πολύ εντάξει. Νόμιζα ότι το, ο σκοπός της έκθεσης είναι να εξετάσει αν μπορεί να γίνει κάτι συμπληρωματικό στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο ο, ίσως πρέπει να προσθεθεί κάτι, να συμπληρωθεί. Και εγώ ευχαρίστως να συνδράμω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν έγγραφα, για παράδειγμα, που έχει καταρτήσει συντάξη κομισιών, μάλλον το 2006 και ο Φιλανδός Πρωθυπουργό κάποια στιγμή εξέτασε τα δυνατά σημεία της Ευρώπης. Πού είναι καλή η Ευρώπη, σε ποιους κλάδους της οικονομίας είναι κορυφαία. Με την έννοια ότι αυτοί οι κλάδοι της οικονομίας βρίσκονται σε αυξανόμενη εξάρτηση από τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τα σχετικά έγγραφα εδώ. Δεύτερον, θεωρώ σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερη σχέση και συνάρτηση με το καθοριστικό σε αυτή τη διαδικασία τον άνθρωπο. Ξέρουμε ότι σε ορισμένους τομείς συρρυκνώνεται η Ευρώπη. Αυτό για τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα. Ήδη στην Κίνα μέσα σε ένα χρόνο εκπαιδεύονται περισσότεροι μηχανικοί τεχνολόγοι, μηχανολόγοι, ε, περισσότεροι από ό,τι στην Ευρώπη σε 10 χρόνια. Οπότε αυτό πρέπει να το δούμε. Με βάση την πολιτική, τη συνθήκη της Λισαβόνας και την πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, βλέπουμε ότι δεν είναι πλήρης η προοπτική για το μέλλον και την πολιτική συνοχή μας θα πρέπει να τη συμπληρώσουμε ακριβώς ως προς αυτό το ελίπον στοιχείο. Επίσης, στις προτάσεις που αναφέρονται εδώ για την περίοδο μετά το 2013, τι προτάσεις υπάρχουν για τις περιφέρειες σύγκλησης, τι προτάσεις συστάσεις για τις άλλες περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια που είναι του στόχου 2 και τι γίνεται με το στόχο 3. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να μιλήσει η πείρα μας τι θα μπορούσε να γίνει εδώ. Ε, χρειάζονται εντατικές διαβουλεύσεις με την Κομισιόν και χρειάζεται και ανταλλαγή γνώσεων στην ε, προπαρασκευαστική ομάδα συζητήθηκε λίγο το μέλλον της πολιτικής συνοχής και συντάχθηκε ένα κείμενο που θα το δούμε άμεσα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής να το δούμε και εμείς. Για το τελευταίο κεφάλαιο, εδώ. Εγώ ευχαρίστως να συνεργαστώ για να καταλήξουμε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, πιο εξειδικευμένες, να δώσουμε προτεραιότητες. Επίσης το συνεκβανόν το εκ των όνου πολιτική για την, πολιτι... την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες, γιατί θα πρέπει να δούμε ευρύτερα το θέμα. Εντάξει, η Ευρώπη, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γύρω μας όμως μεταβάλλεται και ο κόσμος, όπως δείχνουν και οι του ΟΣΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρότερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ μιλώ εξ ονόματος του Ζαν Πολ Πεσέ, ο οποίος νόμιζε ότι θα καθυστερούσε η έκθεση να συζητηθεί και θα έρθει λίγο αργότερα και υπάρχουν ορισμένα σημεία που έχει εκείνος σημειώσει. Πρόκειται για το εξής. Πρώτον, διαπιστώνει ότι η έκθεση αυτή κυρίως βλέπει την υποδομή, τις υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών. Μπορεί αυτό να ισχύει για ορισμένες περιφέρειες, αλλά όχι για την πλειονότητά τους. Νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο ο συνάδελφος Βανίστελ Ρόι. Με βάση την ανάλυση της Ευρώπη 2020 και τη στρατηγική Μπαρόζο βλέπουμε ότι η ανταγωνιστικότητα είναι ευρύτερη αλλά και πιο συγκεκριμένη σε σχέση με επιμέρους τομείς. Καταρχήν μιλάμε για τη γνώση και την καινοτομία. Εδώ έχουμε ένα, μια κεντρική, ε, ένα κεντρικό μέσο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αυτό δεν αναφέρεται εδώ. Επίσης επενδύσεις για αηφόρο ανάπτυξη συγκεκριμένα ε, επηρεάζει την ε, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και όποιος ε, δραστηριοποιηθεί πρώτος σε αυτό το τομέα αυξάνει τις πιθανότητες πώλησης των προϊόντων του στην διεθνή αγορά. Και αυτό λείπει. Η ανταγωνιστικότητα για ε, ορισμένες περιφέρειες μπορεί να έγκυται στην βελτίωση των υποδομών, αλλά δεν είναι πανάκι αυτό το τελευταίο. Η αηφόρος ανάπτυξη και η καινοτομία στα προϊόντα εξασφαλίζουν ε, την ανταγωνιστικότητα, άλλωστε δημιουργούν και θέσεις εργασίας και υπησέρχονται και σε θέματα κοινωνικής συνοχής που σε πιο απομακρυσμένες περιφέρειες με αυτόνομη ανάπτυξη χωρίς εύκολη πρόσβαση και σύνδεση με το κέντρο, ε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό λείπει. Για την παράγραφα 6, να πούμε και κάτι θετικό, συμφωνούμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που παρουσιάζεται εδώ ως δυνατότητα πρόοδου, όμως στην παράγραφο 8 προτείνεται μια, να υπάρξει ένα σύμφωνο μεταξύ Κομισιών, Καρατών Μελών και Περιφερειών, αλλά το 2002 το επιχειρήσαμε αυτό και δεν είχε αποτέλεσμα. Να κάνει λοιπόν ο εισηγητής μια ανάλυση, γιατί δεν λειτουργήσε, όχι να ανατρέξουμε σε αυτή τη λύση η οποία δεν μας πήγε μπροστά τότε. Ε, στην παράγραφο 11 εδώ μπαίνει σε αυτό που συζητούμε τώρα στην ε, ομάδα εργασίας, αναφέρομαι στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κλπ. Εδώ μάλλον δυσκολεύουν τα πράγματα και δεν θα μείνει ως έχει, γιατί τώρα οι συζητήσεις έχουν διευρυνθεί πολύ. Θα καταθέσουμε και σχετικές τροπολογίες, γιατί εξακολουθούμε να είμαστε πεισμένοι ότι ένας συνδυασμός ΑΕΠ βάση συν Gini ε, είναι καλύτερη περιφερειακή πολιτική για το μέλλον, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που δεν ε, καλύπτονται από το κριτήριο 75. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά, Περίμενα με περιέργεια την έκθεση γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα λέει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το περιεχόμενο που συνέταξε ο εισηγητής, αλλά θα ήθελα σε ένα τμήμα, ίσως μπορούμε να προσθέσουμε και ένα μικρό πέμπτο μέρος και να ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό για τη συζητήσεις μας των επομένων μηνών, γιατί η συνοχή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνεισφορά και συμβολή στην ανταγωνιστικότητα. Γιατί υπάρχουν πολλές, πολλοί προβληματισμοί. Έχουμε μητροπόλεις, έχουμε πλούσιες χώρες, αυτό αρκεί για την ανταγωνιστικότητα και δεν χρειάζεται να εφεύρουμε καινούργια πράγματα, κάτι τέτοιο. Ή υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις. Η έκθεση λοιπόν είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για να γίνει αυτή η διευκρίνηση, γιατί χρειάζεται δηλαδή πολιτική συνοχή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ε, ξεκαθαρίσουμε το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, λείπει ένα άλλο κομμάτι, θεωρώ. Όλη αυτή η θεματική για την ε, αηφόρο, η βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι από μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν συνιστά ανταγωνιστικότητα, αλλά χρειάζεται μια κοινή κοινοτική αηφόρος ανάπτυξη ε, ώστε να διασφαλιστεί η διάρκεια της ανταγωνιστικότητας. Μπορούμε λοιπόν κάποια στιγμή να συσκεφθούμε και να δούμε πώς θα τα γράψουμε αυτά με τον καλύτερο τρόπο στην έκθεση, γιατί η έκθεση είναι σημαντική και σε σχέση με αυτά που θα διαπραγματευτούμε και θα συζητήσουμε το φθινόπωρο με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. συγγνώμη. Η κυρία Μανέσκου ζήτησε το λόγο πριν από τον κύριο Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Λουχάν, για το σχέδιο έκθεσης που συνέταξε, γιατί πιστεύω ότι η πολιτική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα είναι δύο παράγοντες κλειδί που συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Και βεβαίως δεν μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικότητα χωρίς μια καλά ανεπτυγμένη πολιτική συνοχής. Γι' αυτό πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να προτείνει πολύ συγκεκριμένες λύσεις και να δώσει πολύ σαφείς κατευθύνσεις όσον αφορά τις ευθύνες που έχουν ε, και θα πρέπει να αναλάβουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, για το κείμενο καθ' αυτό, φυσικά η πολιτική συνοχή υποστηρίζει την ανάπτυξη και επηρεάζει τα πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ε, υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα προβλήματα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η ολοκληρωμένη αντίληψη θα πρέπει να αναφέρεται και να αναπτυχθεί και μέσα στο κείμενο της έκθεσης. Επίσης παρατήρησα ότι το σχέδιο έκθεσης βασίζεται στην ε, σημασία των υποδομών σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Όντως, και οι υποδομές είναι ένα σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι όμως ο μόνος σημαντικός παράγοντας. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, επίσης να λάβουμε υπόψη μας και άλλους τέτοιους παράγοντες όπως η οικονομική μεγέθυνση και η απασχόληση. Σε σχέση με την αύξηση των επιδόσεων των περιφερειών. Και ένας άλλος παράγοντας μπορεί να είναι, η, ο βαθμός απορρόφησης και αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, στο, στην έκθεση αυτή θα έπρεπε να τονίσουμε την σημασία που έχει η ανάπτυξη του επιχειρησιακού δυναμικού ε, της, ε, των, των περιφερειών ε, της επιχειρηματικότητας και επίσης ε, ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει το επιχειρηματικό πνεύμα να ε, αναπτυχθεί σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό να αναπτυχθεί η περιφερειακή και διαπεριφερειακή ανταγωνιστικότητα. Επίσης πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που έχουν τα πιλωτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προσαρμογή στις νέες προκλήσεις και επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθούν οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης για όλα αυτά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμένα η έκθεση με έπεισε Νομίζω ότι έχουμε ένα παράδειγμα εδώ εισηγητή από ένα νέο κράτος μέλος όπου οι ανάγκες είναι διαμορφωμένες διαφορετικό τρόπο. Ε, να πω ε, ότι χωρίς υποδομές, χωρίς ενέργεια, χωρίς επικοινωνιακές υποδομές, χωρίς δρόμους δεν υπάρχει περιφερειακή ανάπτυξη. Στην Ανατολική Ευρώπη έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η βάση. Και μετά Αφού κάνουμε την αρχή, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε και οικολογικά κριτήρια. Στα πλαίσια βέβαια ενός γενικότερου σχεδιασμού. Αλλά είναι πάρα πολύ σωστό να δώσουμε έμφαση στις υποδομές. Και μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες προτάσεις ενδεχομένως. Ίσως ό,τι αφορά τον δίκτυ, αυτό το συντελεστή Gini, το είχα σπουδάσει αυτό όταν ε, μάθαινα γεωγραφία είναι λίγο θεωρητικός. Τι έχει να κάνει σε περιφερειακό επίπεδο η κατανομή του εισοδήματος με την δυναμικότητα μιας περιφέρειας συνολικά. Μόνο το ΑΕΠ μετράει. Όλα τα άλλα νομίζω ότι δεν έχουν τόση σημασία. Οπότε μην τα βάζουμε αυτά. Ε, αλλιώς ε, θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, θα έχουμε ε, ανακατέψει ένα σωρό εταιρών διαφορετικά πράγματα και δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Να ρωτήσω κάτι τον εισηγητή τώρα για τα global grants, αυτές τις ε, παγκόσμιες επιχορηγήσεις ε, στις περιφέρειες η λογοδοσία σε ποιο επίπεδο θα βρίσκεται, γιατί δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποιος θα αναλαμβάνει επί της ουσίας ε, την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη, την δημοσιονομική ευθύνη για την ε, χρησιμοποίηση αυτών των κονδυλίων. Και όταν μιλάμε για διοικητική απλούστευση, νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε ένα μέσον, όπως είπε και η κυρία Μανέσκου, που θα έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πιστοποίηση διοικήσεων, ούτω ώστε να μην γίνεται ξανά και ξανά η ίδια διαδικασία. Αν δείξουμε μια φορά εμπιστοσύνη σε μια διοίκηση, αυτή η εμπιστοσύνη να ισχύει και για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ομιλητής, η κυρία Λούκατς Γεύσκα. Ευχαριστώ. έχω τρεις παρατηρήσεις πολύ συχνά αναφέρθηκε το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ νομίζω ότι το κυρίως θέμα της έκθεσης είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι η εσωτερική ανταγωνιστικότητα. Και στόχος μας είναι να επιτύχουμε παρόμοια ανταγωνιστικότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης, ώστε να βελτιώσουμε τη γενική ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και χαίρομαι που η έκθεση αυτή επικεντρώνεται σε θέματα εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, γιατί άλλη είναι η προοπτική των, χωρών, των νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τελευταίων 10 ή 12 και των χωρών της των 15 αρχικών χωρών μελών. Και χαίρομαι που ο κύριος Λούχαν υιοθετεί και αυτή τη νέα προοπτική. Και ανάλογα με την προοπτική, τα συμπεράσματα είναι διαφορετικά. Πάντως όλοι συμφωνούμε ότι χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς έμφαση στις υποδομές, οι νέες χώρες ε, δεν θα είναι ανταγωνιστικές γιατί χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να καλύψουν το χαμένο έδαφος και να εξισωθούν με τις υπόλοιπες χώρες στην ανταγωνιστικότητά τους. Οπότε αν μείνουν πίσω ορισμένε χώρες δεν θα ε, υλοποιήσουμε το στόχο της ανταγωνιστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης αναφέρθηκε ότι χωρίς επενδύσεις σε μια καινοτόμα οικονομία δεν θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ανταγωνιστική διεθνώς. Συμφωνώ επίσης με τον κύριο Βανίστερ Ρόι που επισήμανε ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που μερικές φορές μας διαφεύγει. Υπάρχει μεγάλη πίεση και μεγάλο άγχος για τους νέους που θέλουν να στραφούν σε τεχνικά επαγγέλματα. Και υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση αυτή εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλε χώρε όπω η Κίνα, η Ινδία. Εκεί οι νέοι κατευθύνονται πολύ περισσότερο σε τέτοια τεχνικά επαγγέλματα. Σε αυτό το θέμα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε αρκετή προσοχή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Matella has also asked for the floor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sigur, voi adăuga câteva lucruri. Unele s-au spus. În primul rând, uh, Aș Προσθέσω και εγώ κάτι. Ελπίζω να μην επαναλάβω αυτά που είπαμε ήδη. Να συγχαρώ τον κύριο Λουχάν καταρχήν για την ε, θαραλέα προσέγγιση του και τον τρόπο ε, με τον οποίο χειρίζεται μια μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στο μέλλον. Νομίζω ότι επουδενή δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να ελαχιστοποιήσουμε το ρόλο της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι μια αρχή ιστορική. Η πολιτική συνοχής κυρίως σκοπό έχει να καταργήσει τις ανισότητες που υπάρχουν, τις ανισορροπίες που υπάρχουν μεταξύ περιφερειών της Ένωσης. Όπως και εγώ, ο κυρίος Λουχάν προέρχεται από μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει πολλά να κάνει σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ο ρόλος των υποδομών είναι σημαντικότατος, όπως ε, άλλωστε πιστεύει και ο κύριος Λουχάν. Οι μεταφορές ε, στις υποδομές είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως για τα καινούρια κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι πικρή ηρωνία να πει κανείς ότι τα ε, αεροπλάνα είναι ο πιο σίγουρος τρόπος σύνδεσης, ε, αλλιώς όταν οδηγεί κανείς η μέση ταχύτητα μειώνεται όσο περισσότερο ανατολικά πηγαίνουμε. Ελπίζω λοιπόν ως κάτοικος ε, ε, σε ανατολική χώρα ότι αυτή η πολιτική συνοχή θα μπορέσει να συμβάλλει στην κατάργηση αυτών των διαφορετικών ε, ρυθμών ανάπτυξης. Επίσης, ένα άλλο θέμα σημαντικό είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων. Και αυτό το καταπιάνεται η έκθεση. Πολύ συχνά πια συζητάμε για περιπτώσεις περιφερειών ή και χωρών που εγκαταλείπουν την ιδέα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων ακριβώς λόγω του, της τρομερής γραφειοκρατίας. Και να σας δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα από μια περιφέρεια της Γαλλίας που το έκανε αυτό. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρούμε αποτελεσματικές, αποδοτικές λύσεις ώστε να διευκολύνουμε τους ετούντες στην πρόσβαση σε κονδύλια. Η έκθεση επίσης μιλάει για την ε, ποικιλομορφία σε περιφερειακό επίπεδο και την εδαφική ανάπτυξη. Εδώ έχουμε νομίζω πολύτιμους πόρους που πρέπει βέβαια να αξιοποιηθούν. Είναι εν πολλής αναξιοποίητοι. Και τέλος θα επαναλάβω πάλι ότι ε, εκτιμώ πολύ την προσέγγιση του εισηγητή στην πολιτική συνοχής και συμμερίζομαι επίσης την άποψή του ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, ανισότητες, ανισορροπίες μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών για να γίνει πιο ομοιογενής η Ευρώπη, εάν θέλουμε να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν είναι κανείς ε, παρόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λουχάνη για τα δικά του σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι σίγουρος ότι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε μια έκθεση πολύ υψηλής ποιότητας σχετικά με το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ όλους για τις ε, παρεμβάσεις σας και για τα σχόλιά σας που πιστεύω ότι είναι επικοδομητικά και απαραίτητα προκειμένου η έκθεση αυτή να γίνει ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Πρώτα απ' όλα για τον τίτλο. Φυσικά ο τίτλος είναι κάπως δύσχριστος, είναι πολύ μεγάλος και αντιστοιχεί σε μια πολύ πλατιά πραγματικότητα και ίσως διαβάζοντας τον τίτλο δεν καταλαβαίνει κανείς τι πρέπει να περιμένει από αυτή την έκθεση. Ο κύριος Βανέσσε Ρόι είπε ότι θα ήθελε να δει πιο συγκεκριμένε προτάσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινητοποιηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι η έκθεση αυτή λέει τι θα πρέπει εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε για να γίνουμε πιο ισχυροί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κύριος Ματούλα είπε ότι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να γίνουμε ισχυροί με την έννοια ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε πρώτα τα δικά μας προβλήματα ε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, οικονομική και κοινωνική, τον οικονομικό και κοινωνικό ανταγωνισμό του υπόλοιπου κόσμου. Και θα το κάνουμε αυτό αν αναπτύξουμε την οικονομία της γνώσης αν επενδύσουμε σε όλες τις κατηγορίες υποδομών και καταργήσουμε τις διαφορές που υπάρχουν σε αυτό το επίπεδο, αν υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για τη δημιουργία ε, μιας πιο δίκαιας ε, αγοράς εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική άνοδο της Κίνας ή της Ινδίας, ο κύριος Βανέσερο είπε ότι μέσα σε ένα χρόνο η Ινδία ε, έχει ε, περισσότερους απόφυτους μηχανικούς από ό,τι έχουμε εμείς μέσα σε 10 χρόνια στην Ευρώπη. Εντάξει λοιπόν, αν ισχύει αυτό, εμείς ε, τι θα κάνουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε 500 εκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν το μισό της Ινδίας. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μην μας ε, ξεφύγουν ε, στον ανταγωνισμό γιατί αυτοί αναπτύσσονται συνεχώς και ίσως σε 5 ή 10 χρόνια αυτοί θα υπαγορεύουν τους όρους ανάπτυξης της ε, παγκόσμια και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, καταπολέμηση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών της. Μιλάμε για τις περιφέρειες της ε, σύγκλησης ή για τη σύγκληση των περιφερειών. Και πρέπει να δεχτούμε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί ιδίω για τα νέα κράτη-μέλη σε σχέση με τους στόχους για τα δυτικά κράτη-μέλη δεν είναι οι ίδιοι. Είναι διαφορετικοί οι στόχοι γιατί έχουμε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Όταν μιλάμε για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως ε, προσθέτουμε αμέσως ότι η διεύρυνση αυτή, η επέκταση, ε, βασίστηκε σε αξίες. Τώρα μιλάμε για οικονομική ανταγωνιστικότητα. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με έρευνα και ανάπτυξη και με την διεύρυνση της αγοράς. Ε, θα πρέπει να βρούμε καλύτερα σχέδια για αυτοαυτοκινητά μας, καλύτερους κινητήρες κλπ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των παγκοσμίων πωλήσεων των αυτοκινήτων μας, ώστε να αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας. Δεν θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ε, Παρ' όλα αυτά, μεταξύ του 2004 και 2007 ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύθηκε κατά 12 κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία ε, ενιαία αγορά, μία εσωτερική αγορά, ε, Έχουμε σχέδια για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς μας. Αυτό έχει και καλά και αρνητικά σημεία. Και τώρα για πρώτη φορά η συνθήκη της Λισαβόνας μας λέει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι θα, δεν θα πρέπει μόνο να μας απασχολεί, ε, ο, να μας απασχολεί ο διαφορετικός βαθμός ανταγωνιστικότητας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί απέναντι στην Κίνα ή στις ΗΠΑ ή τη Ρωσία. Αυτή είναι μια μείζον αλλαγή. Όσον αφορά τώρα την ιδέα να θέσουμε ε, την ανάπτυξη των υποδομών ε, σε ένα κεντρικό σημείο ε, μέσα σε αυτή την έκθεση, φυσικά χωρίς συνοχή στις υποδομές και την πολιτική υποδομών δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική πολιτική συνοχής. Γι' αυτό όντως πρέπει πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα αν ε, θέλουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Υποδομές της τηλεπικοινωνίας, ενέργεια κλπ. Όσον αφορά τώρα τις ε, σχέσεις ανάμεσα στις περιφέρειες στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, πάντοτε λέμε ότι η Ευρώπη του 2020 θα είναι η Ευρώπη των περιφερειών. Βλέπουμε χώρες όπως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, όπου ο καταμερισμός του προϋπολογισμού γίνεται με βάση προγράμματα ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ε, καταπολεμήσουμε, να περιορίσουμε την γραφειοκρατία, να περιορίσουμε, να μειώσουμε τα χρονικά περιθώρια που χρειάζονται για την ανάπτυξη των προγραμμάτων και έτσι να συμβάλλουμε σε μεγαλύτερο βαθμό ανάπτυξης. Επιπλέον πιστεύω ότι εμείς εδώ σε ένα γραφείο στις Βρυξέλλες ή σε ένα γραφείο μιας εθνικής κυβέρνησης σε ένα κράτος μέλος δεν μπορούμε να έχουμε ε, καλή τόσο καλή εικόνα σχετικά με το αναπτυξιακό δυναμικό μιας περιφέρειας όπως έχουν οι ίδιοι εκπρόσωποι της περιφέρειας. και ε, αυτό λέω ότι αν μια κάποια περιφέρεια έχει ε, μια συγκεκριμένη δυναμική, ας εστιάσουμε σε αυτή τη δυναμική και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, Όλοι ξέρουμε ότι η Γερμανία είναι πολύ καλή στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία. Ας υποστηρίξουμε λοιπόν την αυτοκινητοβιομηχανία. Όλοι ξέρουμε ότι η Ανατολική Ευρώπη χρειάζεται καλύτερες υποδομές. Ας εστιάσουμε λοιπόν όντως στην ε, ε, βελτίωση των υποδομών. Όμως, ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς μας. Ε, η κυρία Κράουλ είπε κάτι με το οποίο συμφωνώ. Μίλησε για την αηφορία και όντως θα πρέπει να αποφύγουμε κοντόφθαλμες πολιτικές. Και γι' αυτό ακριβώς αναφέρεται πολλές φορές μέσα στην έκθεση η λέξη συνέχεια. Μιλάμε για την συνέχεια ανάμεσα στους στόχους που θέτουν τα κράτη-μέλη και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια κάποια ε, δομή χρηματοδότησης που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έργα με θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να ε, έχουν μια συνέχεια. Και ε, μιλάω βέβαια για ωφέλη αναπτυξιακά και οικονομικά σε επίπεδο ε, περιφερειών. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα ευρωπαϊκά ταμεία και τη χρήση των κονδυλίων τους μετά το 2013 και γι' αυτό ε, λέω ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πρέπει να είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να την υπόψη. Οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών θα πρέπει να είναι ένα δεύτερο κριτήριο, καθώς επίσης και η ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η πρόθεση μεγάλων πιλωτικών έργων. Όντως, αν θέλουμε να έχουμε ε, σημαντικά αποτελέσματα από οικονομική σκοπιά, θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να ε, κυνηγήσουμε τα μεγάλα έργα, να επιδιώξουμε τα μεγάλα έργα. Όντως, στην έκθεσή μου δεν δίνεται απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε μια απάντηση σχετικά με το ποιος θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Οι εθνικές κυβερνήσει, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να καθοδηγήσουμε ε, το θέμα αυτό και μπορούμε να δώσουμε ε, μια απάντηση με μια πιο ακριβή ε, πολιτική συνοχής, μεγαλύτερη ακριβίας. Ας συζητήσουμε και ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την προώθηση της επιχειρηματικότητας, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα ήταν μάταιο να έχουμε ε, μια ε, σχετικά ε, καλή λειτουργία της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης και διοίκησης αν οι επιχειρηματίες δεν συμμετέχουν, οι επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν και την ιδιαιτερότητα και την δυναμικότητα μιας περιφέρειας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ για την θέση του, γιατί παρόλο που προέρχεται από μια ε, χώρα της Δυτικής Ευρώπης με εξαιρετικές υποδομές, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί αναγνωρίζει την ανάγκη εξισορρόπησης εξίσωσης αν θέλετε, της ποιότητας των υποδομών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θέλουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι αυτό είναι εντελώς απαραίτητο και μιλάω από προσωπική πείρα. Εγώ ε, έτυχε να εργαστώ για μια γερμανική εταιρεία που κάποια στιγμή ε, έψαχνε να βρει νέες ε, επενδυτικές ε, ευκαιρίες και είχε ένα κατάλογο με 30 κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούσε για να επιλέξει τον τόπο της επένδυσης και 20 κριτήρια για τη συγκεκριμένη πόλη μέσα σε αυτή τη χώρα όπου επρόκειτο να επενδύσει. Το δεύτερο από τα κριτήρια ήταν οι υποδομές, η προσβασιμότητα με άλλα λόγια είχαμε ε, καταλήξει σε τρεις ε, ε, επιλογές για τον τόπο της επένδυσης που επρόκειτο να γίνει και ανάμεσα στους τρεις αυτούς επικρατέστερους υποψήφιους επελέγει η χώρα που είχε τις, η περιοχή που είχε τις καλύτερες υποδομές παρόλο που ήταν λιγότερο ανταγωνιστική από άλλες απόψεις. Η επένδυση αυτή ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια που η επένδυση αυτή χάθηκε για τις άλλες δύο πόλεις, για πόλεις επρόκειτο, γιατί ε, δεν είχαν καλές υποδομές, παρόλο που από άλλες απόψεις ήταν ε, καλύτεροι υποψήφοι. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα για να σας ε, δώσω να καταλάβετε πόσο μεγάλη έμφαση δόθηκε στο θέμα των υποδομών, που δημιουργούν μεγαλύτερες ευκαιρίες, ε, μεγαλύτερη δυναμικότητα για μια περιφέρεια και καλύτερες προοπτικές για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την περιφέρεια ή την πόλη. Ποιος θα πρέπει να είναι αρμόδιος, ποιος θα πρέπει να έχει την ευθύνη για τις επενδύσεις. Εγώ έχω το δικό μου όραμα και τις δικές μου απόψεις για το θέμα αυτό. Ας είμαστε ειλικρινείς, είμαστε όλοι προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος αν θέλουμε να συγκρίνουμε τα πολιτικά και διοικητικά συστήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι υπάρχουν τεράστιε διαφορέ μεταξύ του. Είτε μα αρέσει είτε όχι, έτσι έχουν τα πράγματα. Θέλουμε να το συνδυάσουμε αυτό με το θέμα τη ε, πολιτική συνοχή, αυτό είναι ένα άλλο καλό ερώτημα. Πάντω, το πολιτικό σύστημα προβλέπει ότι κάθε τέσσερα χρόνια περίπου πέφτει η προηγούμενη κυβέρνηση και εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση. Αυτά τα κονδύλια, πολλά από αυτά τα κονδύλια, τα διαχειρίζονται ε, κάποιες ε, υπηρεσίες, κάποιες μονάδες ε, και διαχείρισης και το πολιτικό χρώμα κάποιων ε, περιφερειών μπορεί να είναι διαφορετικό ας το πούμε έτσι, από το πολιτικό χρώμα άλλων περιφερειών. Αν συνδέσουμε τις αλλαγές αυτές με τις πολιτικές αλλαγές, ε, με πολιτικά κριτήρια δηλαδή, κάποιες περιφέρειες θα ε, χάσουν γιατί δεν θα έχουν το σωστό πολιτικό χρώμα. Αν λοιπόν δεν ορίσουμε σαφώς που, ποιος έχει την αρμοδιότητα, ποιος έχει την ευθύνη ε, για το σύνολο των περιφερειακών επενδύσεων, Φυσικά πάντα ε, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο θα έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, αυτή την απειλή. Αν το κάνουμε όμως έτσι θα ξέρουμε και θα είμαστε σίγουροι ότι πολιτικοί ή διοικητικοί παράγοντες δεν θα μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονται τα κονδύλια προς τις περιφέρειες. Γιατί μπορεί να έχουμε περιστάσεις, παραδείγματος χάρη, όπου κάποιοι τοπικοί ηγέτες να είναι πιο αποδυναμωμένοι, πιο αδύναμοι, να μην έχουν πολλές ικανότητες, ε, ε, να μην είναι πολύ ικανοί σε κάποια παιδεία. Ε, τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε να υποβαθμιστούν αυτές οι περιφέρειες λόγω της πολιτικής ανικανότητας των ηγετών τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σαφή γραμμή όσον αφορά την γραμμή την αλυσίδα των, της, ε, των αρμοδιοτήτων από την περιφέρεια στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας έχουμε λοιπόν ένα στρατηγικό σχέδιο ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Ας το διαπραγματευτούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί σε επίπεδο Ένωσης έχουμε μια σαφέστερη εικόνα των αναπτυξιακών τάσεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε σαφή κριτήρια ε, για την υποστήριξη της πολιτικής και οικονομικής συνοχής, της δημιουργίας απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ισχυρότεροι από οικονομική σκοπιά και πιο γρήγορα. Και θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε οικονομικά την Κίνα, την ε, Ρωσία, την Ινδία με καλύτερα ε, οικονομικά όπλα η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο μέσα σε αυτή την έκθεση. Είναι κάτι που ακούσαμε από τους ε, παρεμβαίνοντες και συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Ε, έχω ένα οικονομικό background και μπορώ να υποστηρίξω αυτή την ιδέα. Ε, η ανταγωνιστικότητα είναι αυτή που οδηγεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν έρθουν οι περιφέρειες και ο ιδιωτικό τομέας σε θέσεις ανταγωνισμού ένας απέναντι στον άλλον, δεν θα έχουμε δημιουργία ε, θέσεων ενεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν ε, η πολιτική συνοχή να λάβει ένα κεντρικό ρόλο. Πιστεύω ότι υπάρχει δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης για τις περιφέρειες αν εφαρμόσουμε ε, σαφή κριτήρια αν λάβουμε υπόψη μας και τα ισχυρά και τα ε, αδύνατα σημεία κάθε περιφέρειας και αν θέσουμε ένα σαφέστατο στόχο, δηλαδή ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Την Αμερική, την Κίνα, την Ινδία. Και αν θέσουμε και πάλι σαν στόχο ότι αυτό θα πρέπει να το επιτύχουμε το γρηγορότερο δυνατό. Είμαι ανοιχτός ε, σε οποιαδήποτε σχόλια ή τροποποιήσεις θα προταθούν ε, για την έκθεσή μου. Είμαι σίγουρος ότι θα, γίνουν, ε, θα γίνει επικοδομητική συζήτηση για τις τροπολογίες και σας ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά σας. Thank you very much indeed. You have... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναγγείλω την την προθεσμία για τις τροπολογίες που λύγει στις 28 Ιουνίου 12 το μεσημέρι προκειμένου να ψηφίσουμε στις 13 Ιουλίου στην Επιτροπή μας και στη δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ωραία. Επαναρχόμαστε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης γιατί περιμέναμε την εισηγήτρια το θέμα αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση σε σχέση με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διαδικασίες ενίσχυσης και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Μανέσκου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους κοιόδης συζητητές και τους συναδέλφους με τους οποίους συνεννοήθηκα πριν εκπονήσω την έκθεσή μου. Είχα διαβουλεύσεις και με ενώσει τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά όλους όσους με βοήθησαν να καταρτήσω αυτή την έκθεση και να τους διαβεβαιώσω ότι προσπάθησα να λάβω υπόψη τις παρατηρήσεις τους και να συμπεριλάβω όσο το δυνατό περισσότερες ιδέες μπορούσα στην έκθεσή μου. Όπως είπε και προηγουμένως, πιστεύω ότι μια αποτελεσματική πολιτική των ευρωπαϊκών πολιτικών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο χαράζονται αυτές οι πολιτικές, ε, με τον οποίο, τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται, αλλά εξαρτάται η αποτελεσματικότητά τους και από τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής συνοχής και μια ενεργή συμμετοχή της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ακόμη και σε, πρόωρο, σε πολύ προκατακτικό στάδιο του σχεδιασμού αυτής της πολιτικής, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική. Θέλουμε ένα είδος μεικτής επιμερισμένης διακυβέρνησης με τις ευθύνες να αναλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Η ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών αρχών ακόμη σε προνομοθετικό στάδιο είναι πολύ σημαντική, γιατί οι τοπικοί και περιφερειακοί παράγοντες γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου και η συμμετοχή τους από πρώιμο στάδιο εξασφαλίζει μια σωστή πολιτική και πολύ πιο αποτελεσματική. Σε θέματα πολυεπίπεδης διακυβέρνηση θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το οριζόντιο αλλά και το κατακόρυφο επίπεδο. Είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και η συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών φορέων η συνεργασία αυτή μεταξύ όλων των παραγόντων είναι απαραίτητη για μια αποτελεσματική συνεργασία και μια εναρμονισμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επίσης, μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση επιτρέπει την καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η εδαφική συνεργασία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο να παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη που το αμέλησαν μέχρι στιγμής να να υλοποιήσουν τον στόχο των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας και να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της περιφερειακής πολιτικής είναι πολύ πιο αποδοτική και αποτελεσματική για τους δικαιούχους της. Και στο μέλλον πιστεύω ότι αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Από τη στιγμή που τα κράτη-μέλη διαδραμάτισαν κέριο ρόλο στην ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών και τοπικών αρχών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εγώ συνιστώ την ε, ενσωμάτωση στην πολιτική συνοχή μιας τοπικής μεθοδολογίας ανάπτυξης με βάση τις κατατόπους εταιρικές σχέσεις, ιδίως για τα έργα και προγράμματα που σχετίζονται με ζητήματα πόλεων, υπαίθρου αλλά και με διασυνοριακά θέματα. Επίσης χρειαζόμαστε έναν κοινό ορισμό της έννοιας της εταιρική σχέσης και θα ήθελα να παρατηρήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατυπώσει ένα τέτοιο ορισμό. Έτσι θα συγκροτήσουμε γνήσιες εταιρικέ σχέσεις ε, με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Επίσης, ε, απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξακριβώνει με σοβαρότητα την εφαρμογή αυτής της αρχής και να διαδίδει τις βέλτιστες πρακτικές ε, μέσω των εργαλείων της πληροφορικής. Ένα άλλο στοιχείο χρηστής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης εκπορεύεται από τις πρόσφατες αλλαγές του Γενικού Κανονισμού και του Κανονισμού ΦΕΝΤΕΡ είναι σημαντικά όλα αυτά τα βήματα. Η διαδικασία όμως της απλούστευσης θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το 2013. Γιατί ελπίζουμε ότι η κρίση δεν θα διαιωνιστεί και δεν θα πρέπει η απλούστευση να εξυπηρετεί μόνο το στόχο της διεξόδου από την κρίση, αλλά θα πρέπει να έχει και πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Επίσης θα πρέπει να περιορίσουμε την απροθυμία κάποιων τοπικών φορέων και περιφερειακών παραγόντων για την πρόσβαση στα διαφορετικά ταμεία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους δικαιούχους των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά αν θέλουμε μια πολιτική που πραγματικά θα αποφέρει καρπούς, που πραγματικά θα έχει αποτελέσματα, θα εφαρμόζεται εύκολα και θα έχει και πιο ορατά και απτά αποτελέσματα για τους δικαιούχους. Μία τέτοια προσέγγιση θα οδηγήσει και σε μείωση του περιθωρίου λάθους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις επιλέξιμες δαπάνες και τις διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμών. Επίσης είμαι υπέρ των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές, Train the Trainers. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και να ενισχύσει την πρωτοβουλία τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτές στις διάφορες χώρες και θα πρέπει να εξασφαλίσει ανάμειξη των τοπικών και περιφερειακών φορέων σε τέτοια προγράμματα. Επίσης, Είμαι υπέρ της συνέχισης του προγράμματος Έρασμος για τους ε, τοπικούς και περιφερειακούς ε, εκπροσώπους. Και να μην εστιάζεται μόνο αυτό στη διαχείριση των ε, διαρθρωτικών κονδυλίων. Φυσικά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες απαιτούν χρηματοδότηση και μια καλύτερη εταιρική σχέση με την Επιτροπή των Περιφερειών προκειμένου να διευκολυθούν οι επαφές μας με τοπικές και περιφερειακές αρχές. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής, πιστεύω ότι η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής της στρατηγικής του 2020, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών και η αίσθηση ιδιοκτησίας αυτών των πολιτικών από πλευρά τοπικών και περιφερειακών αρχών. Επαναλαμβάνω και πάλι τις ευχαριστίες μου προς τους και ηγετές για τις προτάσεις τους. Φαντάζομαι ότι θα κατατεθούν τροπολογίες από τους συναδέλφους και τις περιμένω με ανυπομονησία για να τις εξετάσω και να τις λάβω υπόψη. Αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Σταυρακάκης έχει μία πρόταση για, τις, ε, για την ε, παράταση του πλαισίου, την διεύρυνση του πλαισίου μάλλον, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο αυτές που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή των Περιφερειών. Και σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι είναι σωστό να μην μιλούμε μόνο για τις 12 νέες χώρες μέλη της Ένωσης. Ο μηχανισμός τεχνικής αρρωγής θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες, και τις παλιές και τις νεότερες. Ευχαριστώ και περιμένω τις παρατηρήσεις Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν σχόλια, παρατηρήσεις. Please. Παρακαλώ. Αφού δεν ζητεί άλλο το λόγο, να ευχαριστήσω θερμά για την καλή συνεργασία. Ήμουν σκιώδης για τους πράσινους. Είχαμε κάνει ε, καλή συζήτηση. Ευχαριστούμε για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης. Είπα στη συζήτηση ότι κάτι που μου φαίνεται κάπως περιοριστικό, όπως, όπως παρουσιάζεται, είναι η κοινωνία των πολιτών και το ζήτημα της διαφάνειας. Θα καταθέσω με κάτι σχετικό. Όμως, κατά τα άλλα, τα σημαντικότερα θέματα τα έχει καταπιαστεί. Α, μια συμπληρωματική ερώτηση, γιατί είπε κάτι για την πιστοποίηση προηγουμένως ο κύριος Πίπερ. Δεν είδα όμως τίποτα για πιστοποίηση στην έκθεσή σας και θα με εξέπλητε αν ε, η Κομισιόν να ε, διαπιστεύσει, να πιστοποιήσει την, ε, του ΣΟΤΑ. Αυτό ως διευκρίνηση. Κατά τα άλλα εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε... Και, ε, Συγχαρητήρια και πάλι στην κυρία Μανέσκου, η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά τονίζοντας τη σημασία της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ως κυρίου παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο και προτείνοντας εφικτούς ε, ε, στόχους όχι μόνο ε, για την προγραμματική περίοδο την επόμενη αλλά και για αυτή. Είναι πάρα πολύ ε, πλήρης, είναι πλήρης η έκθεση, κάνει σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση της ε, διακυβέρνησης και αυτό παίζει κέριο ρόλο για να εξαλειφθούν κάποιες αδυναμίες στην πολιτική αυτή. Δύο σύντομα σχόλια μόνο. Πρώτον, μια μικρή αναφορά στη στρατηγική έκθεση της Κομισιόν για την εφαρμογή των προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής στην περίοδο 2007-2013 θα ήταν χρήσιμη σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να σημειωθεί για παράδειγμα και πάντα σε σχέση με την ανάγκη για την απλούστευση, μπορεί να ε, αναφερθούν τα εμπόδια που εντοπίζουν τα κράτη-μέλη για την γρήγορη υλοποίηση όπως ε, αλλαγές των κανόνων για το δημοσιονομικό έλεγχο και την περιπλοκότητα της διαχείρισης ε, επικαλυπτωμένων ε, προγραμματικών περιόδων κλπ. Και το δεύτερο σχόλιο είναι, θα ζητούσαμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει γιατί σε κάποια κράτη-μέλη παρατηρείται μια μεγάλη αντίσταση στην επίλυση προβλημάτων διοικητικών και προβλημάτων υλοποίησης. Και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η μακρά εμπειρία στην διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Πώς μπορούμε να αντλήσουμε περισσότερα από την ήδη υπάρχουσα εμπειρία. Ευχαριστώ. Mulțumesc. Aș dori să και εγώ θέλω να συγχαρώ τον την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά. Και να την ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε, γιατί και εγώ ήμουν σκιώδης για αυτό το σχέδιο έκθεσης. υπάρχουν κάποια σημεία στην έκθεση αυτή που έχουν τεράστια σημασία. Ένα από αυτά είναι το εξής. Τι θα δώσουμε στους ΟΤΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι ακριβώς θα δώσουμε. Επίσης θέλω να αναφερθώ στο σημείο 17 που αναφέρει την ανάγκη για ε, τυποποιημένους ε, ελέγχους και να ε, θυμίσω ότι είπε ο καθηγητής Μπάχτλερ χθες κατά την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σχετικά με το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, τι ακριβώς, πόσα θα δώσουμε στη, στην τοπική αυτοδιοίκηση αν κάποιος ετών που έχει υποβάλει αίτηση κερδίσει ένα ποσόν από ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο. Θα πρέπει να περάσει από 8 ή 9 διαφορετικές διαδικασίες ελέγχου. Ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου είναι μεγάλη πρόκληση και πρέπει όμως να βρούμε τρόπους για να το πετύχουμε αυτό. Βέβαια, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι σημαντική η έλεγχη. Βεβαίως είναι σημαντικό να υπάρχει έλεγχος και να γίνονται διαδικασίες ε, ελέγχου. Όμως αυτές δεν θα πρέπει να γίνονται εμπόδιο και βάρος για τους ε, δυνητικούς δικαιούχους που πρέπει να ξέρουν ότι όταν κερδίσουν μια χρηματοδότηση θα πρέπει να περάσουν από κάποιες διαδικασίες ελέγχου. Αν μπορέσουμε αυτές τις διαδικασίες ελέγχου να τις βελτιώσουμε χωρίς να υποβαθμίσουμε την αποτελεσματικότητά τους, αυτό θα είναι πολύ καλό. Μια άλλη σημαντική ιδέα που εκφράζεται εδώ στο σχέδιο έκθεσης και που απορρέει από το ευρωβαρόμετρο της Eurostat που λέει σαφώς ότι ο υψηλότερος βαθμός εμπιστοσύνης ε, βρίσκεται σε τοπικούς διοικητικούς φορείς. Το ίδιο βαρόμετρο δείχνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συμμετέχει όσο θα έπρεπε στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Και γι' αυτό στο σημείο 7 στο σχέδιο έκθεσης ε, λέει ότι πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο οι αρμόδιες τοπικές αρχές. Πρέπει λοιπόν να αναθέσουμε, να μεταφέρουμε αρμοδιότητες σε εκείνο το επίπεδο. Πρέπει να γίνει αυτό γιατί είναι φυσιολογικό αυτές οι αρχές να συμμετέχουν περισσότερο και στις διαβουλεύσεις και στις αποφάσεις. Άλλη μια φορά θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε εξαιρετική συνεργασία ε, πάνω σε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο κύριος Ματούλα. Στην παράγραφο 17 γιατί δεν θα μπορούσαμε να πούμε ένα ενιαίο πρότυπο ελέγχου. Γιατί αν ε, μετά από τέσσερα χρόνια δεν υπάρχει εκαθάριση των λογαριασμών, σημαίνει ότι κάτι ε, δεν έχει πάει καλά. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο ελέγχου και αν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπάρχει απάτη, θα πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το κείμενο, το συγκεκριμένο, αλλά καλό είναι να σκεφτούμε και αυτό που είπαμε χθε για την ε, πιστοποίηση και για την ιδέα ε, να υπάρχουν προγράμματα με κοινή ε, διαχείριση. Πράγμα το οποίο θα ισχυροποιήσει την θέση μας. Μιλήσαμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παράλληλα με την πολιτική συνοχής και χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι είναι ανοιχτή στην ιδέα να αξιοποιηθούν κάποια διδάγματα που προέρχονται από την γεωργία. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της περασμένης εβδομάδας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί στόχοι θα πρέπει να συνοδεύονται από στόχους σε επίπεδο κρατών μελών. Αυτή είναι η έννοια της ε, ε πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και επίσης θα μπορούσαμε να βασιστούμε και σε κάποια άλλα σημεία που προέρχονται από αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Συμφωνώ με τον εισηγητή ε, που λέει ότι το πρόγραμμα Έρασμος θα πρέπει να διευρυνθεί. Δεν είχαμε μεγάλη επιτυχία από το πιλωτικό project που εφαρμόστηκε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί κάπως ε, το κείμενο στο σημείο αυτό και στο τέλος στο 10 σχετικά με την ε, ε, συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα από κάτω επίπεδα διακυβέρνησης για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 Αυτό είναι μία από τις βασικές δεσμεύσεις. Για την Κομισιόν ίσως. Αλλά θα πρέπει ε, να δούμε και την εδαφική διάσταση στο σύμφωνο ανάμεσα στις περιφέρειες και τις πόλεις και τους δήμους. Θα πρέπει να δούμε ε, σχετικά με αυτά τα εμβληματικά σημεία τη θέση της Κομισιόν. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Ανδρούλα Ιωάννου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητρία την κυρία Μανέσκου για την έκθεσή της που έχει συγκεκριμένες προτάσεις και θα συμβάλλει στη συνεχή συζήτηση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική συνοχή μετά το 2013. Σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να συζητήσουμε και να προσδιορίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του υποπτικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της, ευθύ, και της ευθύνης εφαρμογής των κρατών μελών. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρθρωτικών έργων και προγραμμάτων. Μα ικανοποιεί η θετική μνήμα που γίνεται στην έκθεση του σχεδίου εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί ο εποπτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά τις αδείξεις ότι το σχέδιο δράση και το ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο για το 2013 βοήθησαν ε, τη διαχείριση και τον έλεγχο, να στραφούν προς σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ με την εισηγητή ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης. Η εγκρίση των εκθέσεων συμμόρφωσης ανα, αναμένεται να ολοκληρωθούν με ελάχιστα προγράμματα να ένα εκκρεμή. Σε ό,τι αφορά το TRE περιφερειών θα συνεργαστεί με την Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού για να μειωθεί το περιθώριο λάθους για τις διαρθρωτικές δράσεις μέχρι το 2012. Επίσης θα γίνουν κάποιες δράσεις μέσω της κοινή στρατηγικής ελέγχου προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία των ελεκτικών αρχών, να εντοπιστούν οι περιοχές ελέγχου να ενισχυθεί η συνεργασία, να αποφευθεί η επικάλυψη ελέγχου και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου αυτού με μια μεγαλύτερη ανάμειξη και ευθύνη των, τοπικών, των εθνικών αρχών. Διοργανώσαμε πολλά σεμινάρια με τις ελεγκτικές αρχές, ιδιαίτερα στα πρώτα επίπεδα ελέγχου που βρίσκονται και τα περισσότερα λάθη. Έγιναν και πολλές τεχνικές συνεδριάσεις με τις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο πρώτου επίπεδου. Εκεί που βρίσκουμε με τα περισσότερα λάθη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά και οι Εθνικές Ελεγκτικές Αρχές. Θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε για την καλύτερη διαχείριση και έλεγχο της τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και μετά από κάποιες καθυστερήσεις θα μπορέσουμε μετά το καλοκαίρι να δώσουμε τις τεχνικές, την τεχνική εροχή που ζητάει η έκθεση και χαιρόμαστε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την παράγραφο 17 και την πρόταση για τον ενιαίο έλεγχο, στον οποίο αναφέρθηκαν και πολλά μέλη της Επιτροπής, ο κανονισμός 2007-2013 αναθέτει πολλές, ελπίδες, ε, πολλές ευθύνες στις ελεκτικές αρχές και εμείς θα ε, στηριχθούμε στις ελεκτικές αρχές. Μάλιστα συστήσαμε μια ομάδα εργασίας που θα συντονίσει τον έλεγχο μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων Διαρθρωτικών Δράσεων ώστε κάθε Γενική Διεύθυνση να αξιοποιήσει το έργο των άλλων. Θα ενισχυθούν οι έλεγχοι λοιπόν και θα πρέπει να αποφευθούν οι επικαλύψεις και με το ελεκτικό συνέδριο, παρόλο που ένα, ένας βαθμός επικαλύψεων θα είναι αναπόφευκτος. Θέλουμε πολιτικές στο μέλλον που θα προσανατολίζονται στα αποτελέσματα. Επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να τηρήσει τις υποχρέσεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Θα πρέπει να ελέγχει την ομιμότητα και την τακτικότητα των διαφόρων συναλλαγών. Θα εξετάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το μηχανισμό εφαρμογής ώστε να μην αποθαρρύνουμε τους επίδοξους δικαιούχους ε, από τη συμμετοχή στα διάφορα έργα και προγράμματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες θα ελέγξει την καλύτερη εφαρμογή των ε, μηχανισμών ελέγχου, πως ζητάει η έκθεση, προκειμένου οι μελλοντικοί κανονισμοί να προσαρμόζονται στις απαιτήσει των προγραμμάτων, στις διαστάσεις των προγραμμάτων, αλλά και στα χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Στην επιμερισμένη αυτή διαχείριση θέλουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα των διαφόρων προγραμμάτων. Αυτό θα είναι σημαντικό στόχο μα και μετά το 2013. Η έκθεση δείχνει ότι αυτά τα τεχνικά θέματα για τη διαχείριση των πολιτικών είναι εξίσου σημαντικά με τους ίδιους τους στόχους πολιτικής. Χαιρόμαστε για την ενεργό ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση και πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα συμβάλλει στις περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κυρία Μανέσκου, για τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους τις υποδείξεις τους και τα καλά τους λόγια για το σχέδιο έκθεσής μου. Εξακολουθώ να είμαι ανοιχτή σε άλλες τροπολογίες, προτάσεις και είμαι πεπισμένη ότι επειδή έχουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα καταλήξουμε σε μια έκθεση η οποία θα δίνει συγκεκριμένες λύσεις σε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Αναφέρομαι στην απλούστευση τους ελέγχους, την συνεργασία των τοπικών περιφερειακών αρχών, πραγματική συμμετοχή των αρχών αυτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην προνομοθετική διαδικασία. Επίσης να επαναλάβω την ανάγκη για αυξημένη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της τεχνικής υποστήριξης. Μιλώ για υποστήριξη ε, των περιφερειακών και τοπικών αρχών μέσα από την ε, τεχνική υποστήριξη. Επίσης υπάρχει ανάγκη για πιο στενή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εποπτεία. Και ελπίζω ότι στο τέλος όχι μόνο θα έχουμε καλύτερη έκθεση, αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εις ό,τι αφορά την πρόσβαση των περιφερειακών και τοπικών αρχών στα ευρωπαϊκά κονδύλια και φυσικά καλύτερη πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Και πάλι σας ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι η 1η Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα γίνει 27-28 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια θα πάει το θέμα τον Οκτώβριο στο Στρασβούργο. Τώρα, προχωρούμε στο σημείο 11 που είναι η γνωμοδότησή μου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες προκλήσεις. Η κυρία Μπέργκερ. You want to take the floor. Yes. Κυρία Μπέρντερ, ζητείτε το λόγο. Ναι. Χαιρετίζω την ευκαιρία να ξαναδούμε αυτό το περίπλοκο θέμα και τις προσπάθειές μας σχεδιασμού για τις ε, θαλάσσιες παράκτιες περιοχές. Ευχαριστούμε και για την γνωμοδότηση. Όμως η έκθεσή σας δεν είναι τόσο ισορροπημένη, ισόρροπη όσο θα ήθελα. Επικεντρώνεται στα νησιά κυρίως. Πρέπει... Ε, ε, ε, και ε, να ξέρουμε τι είναι τα νησιά και εμεί θεωρούμε ότι είμαστε νησί. Βέβαια εσεί αναφέρεστε σε νησιά μικρότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Θα συμπεριλάβω τροπολογίε ε, για τους εξής τομείς προστασία θαλασσίων, συστημάτων, οικοσυστημάτων, τον τουρισμό, παράκτια παρακολούθηση, περιπολίες. Τώρα, Εν ώψη της κλιματικής αλλαγής δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα, πώς θα βοηθηθούν τα οικοσυστήματα. Ήδη παρατηρούμε αλλαγές με θύελες, καταιγίδε, πλημμύρε, ε, θέρμανση, αυξήση της θερμοκρασίας των θαλασσών κλπ. Είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε και οι προειδοποίησεις. Κάποιοι λένε ότι θα αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας, άλλοι λένε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις δυτικές ακτές. Ε, ακούμε ότι το ρεύμα του κόλπου θα αλλάξει, οπότε θα γίνουν ψυχρότερες οι θάλασσες και θα έχουμε τύπου, ε, χειμώνες αρκτικού τύπου και αυξημένη ποσότητα άλατος στις θάλασσες. Όλα αυτά επηρεάζουν πολύ τα οικοσυστήματα που τα, έτσι όπως τα ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ε, προστατευτικές νομοθεσίες για την προστασία ε, για τα πουλιά, οι οδηγίες ε, μέχρι εκπομπές άνθρακα από τα μεγάλα πλοία. Η Natura 2000 και άλλα οδήγησαν σε πληθώρα ε, προστασίας ε, και ταξινόμησης ε, των ακτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε έξι διαφορετικά είδη προστασίας και αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε για να διευκολύνουμε την κατανόηση της προστασίας και τι ισχύει για τα οικοσυστήματα των ακτών μας. Οι παράκτιες περιοχές, περιφέρειες επίσης είναι πολύ σημαντικές. Ε, μπορεί να έχουμε καλύτερη παραγωγή ενέργειας, ε, αιωλική ενέργεια, ενέργεια από τα κύματα, ε, την παλήρια. Όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού που θα λάβει χώρα και σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διακινούνται ναύλοι κλπ. Στις παράκτιες περιοχές το εμπόριο και ο τουρισμός. Στη δική μου την περιφέρεια που είναι η πιο κοντινή στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι το Ντόβερ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός λιμίν για το ευρωπαϊκό εμπόριο, 80 ε, δις στερλίνες είναι ο τζίρος εκεί και πολλοί μεταφορείς το χρησιμοποιούν. Έχουν διπλασιαστεί 2,5 εκατομμύρια ε, μεταφορείς το μεταφορικές μονάδες περνούν από εκεί. Ε, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας την ομαλή ε, εργασία και την αποφυγή ε, εργασιακών ε, απεργιών κλπ. Επίσης ε, είναι πολύ σημαντικό και για τη διέλευση των τουριστών. Είναι εκατομμύρια που περνούν από το λιμάνι αυτό. Και εσείς αναφέρεστε σε αυτό το θέμα. Όμως ε, είναι τεράστιος ο όγκος των τουριστών που περνούν τη μάγχη. Επίσης 4 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποιούν ετησίω το λιμάνι του Ντόβερ. Το Ντόβερ λοιπόν είναι ένα λιμάνι βέβαια, αλλά είναι τεράστια η διακίνηση από εκεί και 80% πάει προς το καλέ. Σε μια περιοχή που από άποψη ναυτιλίας ε, είναι από τις πιο σημαντικές για την ε, κίνηση από βοράν προς νότον. Είναι λοιπόν πολύ ε, μεγάλη κίνηση σε αυτή την θαλάσσια οδό. Ε, εσείς επίσης αναφέρεστε σε κάτι που ίσως πρέπει να διευκρινιστεί, δηλαδή όταν αναφέρεστε σε μικρές αποστάσεις ε, νομίζω ότι η Επίτροπος Δαμανάκη ήδη δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα για να δει πώς θα επιδράσει η πολιτική, κοινή πολιτική για την αλία όλα αυτά. Εσείς αναφερθήκατε στις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Ε, πρέπει λοιπόν να δούμε ε, και το ζήτημα της περιπολίας παράκτιων ε, περιοχών και ε, αν δεν έχει πιστεί για την ανάγκη θα πρέπει να δει τα στοιχεία για την, το λαθρεμπόριο και κοντραμπάντο που λαμβάνουν χώρα εκεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει συνεργασία ε, όλων των αρχών για την προστασία των παράκτιων περιοχών. Ε, αυτή είναι μια συνεργασία μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών και θα πρέπει να υπάρχει μια, ε, ένα συντονισμός μεταξύ των αρχών γιατί είναι περίπλοκο το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά η συνεργασία μου μαζί σας πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κεντέκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τομέα που μου είναι πολύ προσφυλής όπως το ξέρετε, είναι η αλία. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην αλία στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πολιτική της αυτή επιμένει στις συνέργειες ανάμεσα στο τομέα σε τομείς και τομεακέ πολιτικές που σχετίζονται με τη θάλασσα. Η Αλία έχει ένα κεντρικό ρόλο ε, στα πλαίσια αυτά και για τις παράκτιες περιοχές βέβαια και η ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έχει σκοπό τη μαγιστοποίηση της ανάπτυξης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψη της η πολιτική αυτή του, το ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αλίας και της ε, ε, σε σχέση με την διατήρηση των αλληλευτικών αποθεμάτων και την πρόθεση ερευνητικών προγραμμάτων. Από αυτή την άποψη, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας είναι εντελώς απαραίτητη για να καταλήξουμε σε μια αηφόρο διαχείριση και πιο αποτελεσματική διαχείριση των ε, θαλάσσιων και παράκτιων πόρων ε, Επίσης είναι επιθυμητό να θεσπιστούν μηχανισμοί διαβούλευσης για την ε, ε, λήψη των αποφάσεων στο επίπεδο της ε, κοινή ελευθερικής πολιτικής και της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Και θα πρέπει να υπάρχουν μεικτά όργανα διαβούλευσης όπου θα, συ, συγκεντρώνονται εκπρόσωποι και της αλίας και της συναυτιλίας για να αναπτυχθεί ένας διάλογος μεταξύ τους. Χρειάζεται μια ε, οριζόντια πολιτική, μια ολοκληρωμένη πολιτική που δεν θα πρέπει να ξεχνάει τη διασφάλιση μιας ε, βιώσιμης αλίας, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον βέβαια, που είναι πηγή οικονομικής ευημερίας για όλους τους εμπλεκόμενους. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και να επαγρυπνούμε για αυτή τη διάσταση στα πλαίσια της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκτιμώντας προφανώς την ε, δουλειά που κάνατε, ε, θα ήθελα ωστόσο να σημειώσω ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με το θέμα που συζητάμε και το γενικότερο πλαίσιο της έκθεσης που καλούμαστε να εξετάσουμε και να ψηφίσουμε. Το πρώτο και το πιο σημαντικό που θα ήθελα να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, είναι το γεγονό ότι η πολιτική θαλασσών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ολοκληρωμένη όπω ονομάστηκε, στην ουσία καλύτερα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τον ε, του μεγάλου κεφαλαίου, του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου, στον ανταγωνισμό με τους ανταγωνιστές στις παγκόσμιες αγορές και αυτό ε, με κόστος στις συνθήκες εργασίας των αυτεργατών, το περιβάλλον και αν θέλετε ακόμα και τις συνθήκες ανάπτυξης ε, των οικονομιών των χωρών μας. Ε, σε σχέση με αυτό θα ήθελα να σας σημειώσω ότι μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην έκθεσή σας στην ανάγκη παραδείγματος χάρη να μην υπάρχει περαιτέρω απελευθέρωση του καμποτάζ και εννοώ ε, περαιτέρω απελευθέρωση του, του καμποτάζ σε πληρώματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γνωρίζετε, αυτό ήδη υπάρχει, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά υπάρχουν τώρα πιέσει αυτή η απελευθέρωση να γίνει και για, για πληρώματα εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σημειώνουμε αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε, γιατί ήδη στην έκθεση, την αρχική έκθεση, Δυστυχώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην ανάγκη εκπαίδευση των ναυτικών, παρά μόνο στην ανάγκη εκπαίδευση των ε, αξιωματικών του εμπορικού ε, ναυτικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκε πραγματικά γαλέρα στα πλοία τη ε, ναυτιλία, κάτι που έχει βεβαίω συνέπειε και για την ασφάλεια των επιβατών και για, την, και για τα ζητήματα τη προστασία του περιβάλλοντο. Άρα ένα ζήτημα σημαντικό πρέπει να είναι το θέμα του καποτάζ. Δεύτερο ζήτημα σημαντικό ε, ξέρετε πάρα πολύ καλά το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας και φαντάζομαι και αλλού ε, με, την, ε, με τους νόμους της αγοράς και που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά νησιά να μένουν αποκομμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα από την υπόλοιπη χώρα, βδομάδες, μήνες, μέρες, είτε γιατί οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλέ και δεν μπορούν οι φτωχοί άνθρωποι να επικοινωνούν, είτε γιατί δεν είναι κερδοφόρες οι γραμμές και δεν υπάρχουν πλοία, πάρα πολύ απλά. Και έτσι ε, ο καθένα σα λύσει το πρόβλημά του όπως μπορεί με τεράστιε συνέπειε από κάθε άποψη. Σε συνθήκε δε όξυνση τη οικονομική κρίση, διότι αυτό ε, περιμένουμε ακόμα αν θέλετε και ασθενού ανάπτυξη. αυτά τα προβλήματα θα γίνουν ακόμα πιο έντονα από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν μέτρα, αν και εμεί είμαστε αρκετά και εξαιρετικά απεσιόδοξοι. Τρίτο ζήτημα, προστασία του περιβάλλοντο. Διαβάζω και ακούω ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις για, τις, ε, ε, για την εξόριξη πετρελαίου στις θαλάσσιες πλατφόρμες, στις ευρωπαϊκές θαλάσσιες, είναι πολύ πιο αυστηροί από ό,τι είναι οι όροι στις ΗΠΑ και από ό,τι είναι ε, η περίπτωση της BP στο κόλπο του Μεξικού. Όμως, πρέπει να σας πω κύριε Πρόεδρε, ότι μετά για τα τελευταία γεγονότα είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για το τι μας περιμένει. Δεν έχω φυσικά καμία ψευδέστηση ότι μπροστά στο κέρδος και μάλιστα στο μεγάλο κέρδος και στο μονοπωλιακό κέρδος δεν έχουμε παρόμοιες καταστάσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι σχεδόν σίγουρο γι' αυτό. Εξάλλου η BP είναι βρετανική εταιρεία, άρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι. Όμως μετά και από αυτό το γεγονός κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνετε. Κάτι πρέπει να ε, μας προβληματίσει και να προχωρήσουμε. Τέλος, ανεμογεννήτριες, πράσινη ανάπτυξη και τα γνωστά. Θα ήθελα να σημειώσω καταρχήν για να μην υπάρχουν και αυταπάτες ότι ναι μεν χρειάζεται μια πράσινη ανάπτυξη διότι η κατάσταση του περιβάλλοντος είναι απαράδεκτη όμως όσο καιρό αυτά τα μέτρα είναι στα πλαίσια του καπιταλιστικού κέρδους και των μονοπωλίων δεν θα έχουμε σημαντική βελτίωση αν θέλετε μπορεί να έχουμε βελτίωση σε έναν τομέα και χειροτέρευση στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει είναι σοβαρό το ζήτημα με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε θαλάσσιες παράκτιες περιοχές που όπως γνωρίζετε προκαλούν πολύ σοβαρά προβλήματα και κατά τη γνώμη μου, ε, τουλάχιστον στη χώρα μου, αγνοούνται επιδεκτικά και παντελώς οι γνώμες των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να εγκατασταθούν ε, μεγάλες ήδη εγκαταστάσεις στη θάλασσα που προκαλούν πολύ σοβαρά ε, προβλήματα. Προφανώς κοιτασόμαστε υπέρ των ήπιων μορφών ενέργειας, δεν χωράει καμία αμφιβολία στο ζήτημα αυτό, όμως δεν μπορεί και αυτό το ζήτημα να υποτάσσεται στο ε, καπιταλιστικό κέρδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αγκουράκη για τις παρατηρήσεις σας. Απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήταν μια γνωμάτιση και όχι ένα report και γι' αυτό εστιάστηκε ακριβώς σε ορισμένα σημεία. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Mr. Ponga, the floor is yours. Merci, Monsieur Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή, το συντάκτη της γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση και να πω σήμερα ότι το οικονομικό κόστος εξαιτίας έλλειψη συντονισμού δείχνει πόσο σημαντική είναι μια ολοκληρωμένη ακριβώς θαλάσσια πολιτική. Η εφαρμογή μιας τέτοιας ολοκληρωμένης πολιτικής ε, θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και σε υφόρο καινοτομία για τις ε, θαλάσσιες περιοχές. Και μάλιστα πολλέ ε, ευρωπαϊκέ περιφέρειε αναγνώρισαν την σημασία του τομέα και αφιέρωσαν αρκετά κονδύλια προκειμένου να ενισχύσουν το δυναμικό του και να το αναδείξουν. Αυτό μα είπε χθε και ο συντάκτη τη γνωμοδότηση και αυτό έγινε στην Γαλλία με τη Βρετάνη. Για την περιφέρεια αυτή μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική θα οδηγεί στην ανάπτυξη των ακτών, στον αηφόρο τουρισμό, αλλά και σε ένα καλύτερο θαλάσσιο σχεδιασμό με περιφερειακή βάση μια τέτοια περιφερική δράση θα πρέπει να έχει και ευρωπαϊκή διάσταση και πιστεύω ότι η έννοια της εδαφικής συνοχής είναι θεμελιώδου σημασία για να αντιληφθούμε και να βελτιώσουμε το συντονισμό στη χρήση των θαλασσών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Επίσης, υπεραπόμακρες περιοχές ενδιαφέρονται και θίγονται ιδιαίτερα από το πρόβλημα των μεταφορών και το 95% των εμπορευμάτων προς την ε, υπηρετική Ευρώπη γίνεται μέσω θαλασσών. Οπότε θα πρέπει να ενισχύσουμε τις αναπτυξιακές στρατηγικές που θα προσαρμόζονται όμως στον υπεραπόμακρο χαρακτήρα αυτών των περιοχών και στην εξάρτηση που έχουν. Ευχαριστώ, επαναλαμβάνω και πάλι το συντάκτη για την γνωμοδότησή του. Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω και κάποιε τροπολογίε με το περιεχόμενο που προανέφερα. Ευχαριστώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, προφανώς έχουμε μια βάση για να προσθέσουμε ζητήματα, μια καλή βάση και εννοώ το σχέδιο γνωμοδότησης του κύριου Σταυρακάκη εκ μέρους της Επιτροπής μας ε, όμως ε, μια πρώτη ανάγνωση του σχεδίου έκθεσης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική ε, από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ε, μας υποχρεώνει να προσθέσουμε κάποια ζητήματα πολύ σύντομα τα οποία και θα κάνουμε πιο συγκεκριμένα με τροπολογίες στη συνέχεια. Το πρώτο που κάνει εντύπωση γιατί ζούμε την εποχή της κλιματικής αλλαγής ότι υπάρχει πολύ ανεπαρκής αναφορά και στα δύο κείμενα ε, στον ρόλο που θα πρέπει να παίξει η ναυτιλία στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο σχέδιο έκθεσης, κάπου στο τέλος, υπάρχει μια αναφορά στη Λευκή Βίβλο για την κλιματική αλλαγή, αλλά τίποτε παραπέρα. Ε, στο σχέδιο γνωμοδότησης λοιπόν της Επιτροπής μας θα πρέπει να γίνει αναφορά σε αυτή την ε, έλλειψη. Και θα θέλαμε να δούμε πιο συγκεκριμένες ε, προτάσεις, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με τις ε, συνδυασμένες μεταφορές ή τη μετάβαση από χερσαίες σε θαλάσσιες μεταφορές ή την ε, σιδηροδρομική διασύνδεση των λιμανιών για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές. Σε κάποια λιμάνια, επειδή πρέπει κανείς να σημειώσει ή είναι ε, απλώς ανεπαρκείς οι άνθρωποι ή και κάποια συμφέροντα δεν έχουν ε, ευνοήσει την ε, σιδηροδρομική διασύνδεση και αυτό είναι απαράδεκτο. Ε, το λέμε λοιπόν και από άψη των μεταφορών ως επιχείρημα και από την άποψη ε, της ε, εξυπηρέτησης της διακίνησης αγαθών και τελικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα θέλαμε επίσης να ε, δούμε μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων από το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να υπάρχει και μεγαλύτερη μέρημνα στον σχεδιασμό των ε, παράκτιων εγκαταστάσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κλιματικές αλλαγές στα επόμενα χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί περισσότερο ο χωρικός σχεδιασμός και γι' αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην ε, προσέγγιση των οικοσυστημάτων, να ενσωματώσει περισσότερο τους στόχους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κυρίως για την προστασία των πτηνών και των οικοτόπων, αλλά και την οδηγία πλαίσιο για το νερό. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στον χωρικό σχεδιασμό καλές πρακτικές, αλλά και να γίνει εκτεταμένη χρήση των τεχνικών εκτίμησης επιπτώσεων στο παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την ε, Επιτροπή μας, θα πρότεινα να κάνει την πρόταση για ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για τις μακροπεριφέρειες, όπως η στρατηγική του Δούναβη ή ακόμα και μια αντίστοιχη για τη Μεσόγειο, όπου υπάρχει ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεμόπουλε. Οι παρατηρήσεις σας ήταν χρήσιμες πραγματικά και ε, θα μας δοθεί ευκαιρία να συνεργαστούμε πολύ στενά. At this point I'd like to give the floor to Mr. Van Nistelrooy. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Φαν Νίστελρόι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να επενέσω τον εισηγητή για τη σύντομη και καλή έκθεση. Δύο πράγματα δίνω ε, στροφή για σκέψη που αφορά και τις συζητήσει στην Επιτροπή μας. Καταρχήν, η εδαφική διάσταση της περιφερειακής πολιτικής, γιατί η Κομισιόν τώρα επεξεργάζεται μία στρατηγική. Ε, περιμένω Περιμένω, περιμένω μέχρι να έχω την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν λοιπόν τώρα επεξεργάζεται μια στρατηγική για τους μακροκανόνες και εκεί στηρίχθηκε η ιδέα μιας πρωτοβουλίας για την ακτή του Ατλαντικού. Ξέρετε τη θέση μας εδώ. Είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί εις ό,τι αφορά τους ε, μακροκανόνες. Ε, δεν θέλουμε αυξημένη γραφειοκρατία και αυξημένα κονδύλια. Αλλά καλό θα ήταν να αναπτύξει η Επιτροπή μας μια τέτοια πρωτοβουλία. Ξέρω το CPMR, την οργάνωση των περιφερειακών θαλάσσιων περιοχών και ξέρω ότι έχει ο οργανισμός αυτός αναπτύξει κάτι και αναφέρεται και στις μακροπεριφέρειες. Αυτό θα τέριαζε και με το στόχο 3 του κανονισμού για τη συνοχή. Το τρίτο μέρος του γενικού κανονισμού εννοώ. Τώρα, αν το δούμε διεξοδικότερα το θέμα αυτό, θα μπορούσε να γίνει και στις άκρως απομακρυσμένες περιοχές. Αν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα με την πολιτική μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τη Βαλτική, το Δούναβι, τις ακτές του Ατλαντικού. Γιατί να μην βάλουμε μέσα και τις εξόχως απόκεντρες θαλάσσιες περιοχές. Τότε θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο πλαίσιο αναφοράς ώστε οι περιφερειακή πολιτική να ασχοληθεί ειδικά με την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Ίσως κάποια στιγμή με την ησυχία μας θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε το θέμα και να δούμε μήπως ε, ε, και αν θα υποβάλει την πρωτοβουλία της τον Οκτώβριο Κομισιόν. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Έντι Χάρντοκ από την Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που άργησα λιγάκι. Καλωσορίζω τα σχόλια που έγιναν. Πρώτα απ' όλα αυτό που έχετε μπροστά σας είναι τέσσερα έγγραφα από την Κομισιόν που αρχίζει να παγιώνει τη δουλειά που ε, ξεκίνησε το 2006 μέσω της ε, δημοσιονομικής ε, βοήθειας που μας έδωσε το Κοινοβούλιο και για την οποία είμαστε ευγνώμονε. Έχουμε και την έκθεση πρόοδου, την οποία δεν θα αναπτύξω. Έχουμε πολύ ε, ε, δραστήρια συνεργασία με, το, με τις διάφορες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμείς, σαν δημόσια υπηρεσία, είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη, για τη συνεργασία. Νομίζω ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα δείχνει την ε, σημασία της ανάπτυξης αυτής της πολιτικής. Καλωσορίζουμε την έκθεση της κυρίας Μάης που συζητάται στην Επιτροπή Τραν, καθώς επίσης και ε, την ε, ε, γνωμοδότηση του κυρίου Σταυρακάκη και βέβαια και ο ρόλος του Intergroup είναι πολύ σημαντικός. Επίσης βλέπουμε ότι αυτή η συνοπτική ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, είναι πολύ σημαντική για να γιατί υπάρχει μια έντονη, μια στενή σχέση ανάμεσα στην ε, ε, πολιτική συνοχή και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και επίσης η συζήτηση που γίνεται σήμερα δείχνει τη στενή σχέση ανάμεσα σε αυτές δύο πολιτικές. Μπροστά σας έχετε την συζήτηση για αυτές τις τέσσερις ειδικές εκθέσεις που έχει η κομισιόν, ε, μεταξύ των οποίων και αυτή για τη Μεσόγειο, καθώς επίσης έχουμε και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη, ε, πολύ σύντομα όπως υποσχέθηκε, θα υποβάλει μια έκθεση, θα κάνει μια ανακοίνωση για το επιστημονικό κομμάτι ε, της θαλάσσιας πολιτικής, ε, ε, τις κλιματικές αλλαγές επίσης. Επίσης, ε, ε, θα έχουμε για κάποια γεωγραφικά έγγραφα ε, για τις μακροπεριφέρειες ή οτιδήποτε άλλες μορφές θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Το γεγονός όμως ότι θα πρέπει να έχουμε ένα συνεκτικό γεωγραφικά έγγραφο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να κάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις για πολιτικές. Ε, ε, επίσης η κυρία Δαμανάκη αναφέρθηκε στο γεγονός ότι έχουμε πρόθεση να κάνουμε κάτι και για τον Ατλαντικό. Ε, την περασμένη εβδομάδα έγινε μια αποκαλή, πολύ καλή διάσκεψη με το ΣΥΠΙΑ ΡΕΝ στην ΡΕΝ. Δεν βρισκόμαστε λοιπόν σε θέση απομονωμένη στην Κομισιόν. Ε, συνεργαζόμαστε με όλους τους εμπλεκόμενους και με τα κράτη-μέλη. Ε, ξέρω βέβαια ότι μιλάω στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν ε, στο όλο αυτό εγχείρημα. Φυσικά οι ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες έχουν το ρόλο να παίξουν σε αυτό το πλαίσιο Αναφερόμαστε στις περιφέρειες αυτές σαν ένα μπλοκ που είναι σωστό βέβαια για διάφορες πολιτικές, αλλά αν το δούμε γεωγραφικά, έχει περισσότερο νόημα οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές να ενσωματωθούν στις περιοχές όπου ανήκουν. η Γουιάννα, Μαρτινίκη, η Γουαδελούπη, παραδείγματο χάρη, δεν ανήκουν περισσότερο τόσο στον Ανατολικό όσο στην Καραϊβική ναι λοιπόν, από μια μεριά να δούμε σαν ένα σύνολο τις άκρως αποκλεισμένες περιφέρειες, αλλά να δούμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ε, και να τις τοποθετήσουμε στο συγκεκριμένο πλαίσιο όπου ανήκουν. Ε, αυτή είναι μια γενική παρέμβαση λοιπόν μια, που ήθελα να κάνω στη σύντομη παρέμβασή μου. Θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω ε, εκ μέρους της Κομισιόν για την υποστήριξή σας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που ξεκίνησε δειλά-δειλά αλλά οριμάζει πλέον και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα χρήματα που μας δώσατε σαν Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη πιλωτικών προγραμμάτων. Ε, τα χρήματα υποστηρίζουν τις πολιτικές και όχι το αντίθετο. Ε, για να μπορέσουμε όμως να συνεχίσουμε θα ε, χρειαστούμε κατά πάσα πιθανότητα κάποιο επίπεδο χρηματοδότησης για τα επόμενα τρία χρόνια. Όλα αυτά θα έρθουν λοιπόν στο επίπεδο του Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξή σας και για τα επόμενα τρία χρόνια των δημοσιομικών προοπτικών. Ευχαριστώ. Thank you very much Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω και πάλι θερμά την κυρία Καρτίν Μπέρντερ, τη Σκιώδη Ηγήτρια και όλους όσους υπέβαλαν πολύ επικοδομητικά σχόλια και παρατηρήσεις. Περιμένω ανυπόμονα τις τροπολογίες σας. Η, τροπολογική η προθεσμία για τις τροπολογίες λίγη στις 28 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι, προκειμένου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 13 Ιουλίου και στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου, στη δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ. Με βάση το άρθρο 49 θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, οι θα αφορούν μόνο τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ε, και σε αυτό το πλαίσιο συνέταξε εγώ τη γνωμοδότησή μου. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο της της διάταξης, το 12, που αφορά την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαίσιο για την έρευνα. Το λόγιο ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ. Αρμόδια κατ' ουσία για την έκθεση αυτή είναι η Ήτρε. Είναι έκθεση πρωτοβουλία για την απλούστευση το, της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαίσιο για την έρευνα. Και μάλιστα στις 30 Σεπτεμβρίου θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή στην ε, Επιτροπή Βιομηχανίας ε, και έχει μεγάλη σημασία εν ώψη του επόμενου Υπουργικού Συμβουλίου για την έρευνα και την καινοτομία που θα γίνει τον Οκτώβριο. Ε, η Επιτροπή μας θα γνωμοδοτήσει επί της εκθέσεως θα ψηφίσουμε στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ θα εξετάσουμε τον Ιούλιο την γνωμοδότηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ολοκληρώσει την εκπόνηση της γνωμοδότησης. Θα σας την υποβάλω στις βραχές προθεσμίες που με δεσμεύουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και σε όσο περισσότερες μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση για την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαίσιο έρευνας. Και στην ανακοίνωση αυτή υπενθυμίζει τη σημασία της ε, έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, να ανακτήσουμε ε, την οικονομική ανάπτυξη, να την προστατεύσουμε και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Φυσικά η πολιτική συνοχή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των, ε, του δυναμικού καινοτομία των περιφερειακών οικονομιών και της συμβολής τους στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά εργαλεία και μηχανισμούς για να ενθαρρύνει την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, πρώτα απ' όλα το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη με πάνω από 50 δις ευρώ το αφιερώνει στη θεμελιώδη έρευνα και τη τεχνολογική ανάπτυξη για την επταετία 2007-2013. Βέβαια, η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού αυτού είναι περιορισμένη εξαιτία τη περιπλοκότητα εφαρμογή του. Γιατί οι διαδικασίε είναι χρονοβόρε, περίπλοκε ε, ε, και δεν συνάδουμε τους στόχους έρευνας και την ανάγκη ελαστικότητας προκειμένου να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει πολλές τεχνικές απλουστεύσεις στο πρόγραμμα πλαίσιο, για παράδειγμα τη βελτίωση της προκήρυξης την υποβολή προσφορών, ενοποίηση των λογιστικών μεθόδων μεταξύ της Ευρωπαϊκής και Εθνικής Χρηματοδότησης, η προσφυγή στις μεθόδους του μέσου κόστους για να μην γίνεται ξεχωριστή η συμπερίληψη κάθε ξεχωριστού κόστους και επίσης ανατολισμός προς την επίτευξη αποτελεσμάτων. Έτσι απλουστεύονται οι διαδικασίες εφαρμογής στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει και μια καλύτερη διευκρίνηση του προγράμματος αυτού σε πολύ πρώιμο στάδιο. Ο κύριος Λάμπερτ Βανίστελ Ρόι σε σχετική έκθεση τόνισε την ανάγκη αναζήτηση συνεργειών μεταξύ των διαφόρων ε, κοινοτικών μηχανισμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνοχή στι κοινοτικέ δράσει μεταξύ του 7ου Ερευνητικού Προγράμματο Πλαισίου, των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Προγράμματο Πλαισίου για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα. Συμφωνώ με τι συστάσει τη έκθεση Βανίλστερ Ρόι και στην γνωμοδότησή μου θα επισημάνω ότι χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των ερευνητικών ε, προγραμμάτων που έχουμε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητά του. Επίση, θα επιμείνω στην εδαφική διάσταση του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου. Χρειαζόμαστε διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και θα πρέπει να την εθαρρύνουμε στα ερευνητικά προγράμματα. Επίση θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρο στην ανάγκη τη ε, ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Συνοχής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ε, καινοτόμε δράσεις. Θα προτείνω κάποιε συστάσει για τη διακυβέρνηση του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου. Το περιφερειακό επίπεδο, κατά τη γνώμη, είναι το δέον επίπεδο για να τονώσουμε την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τι ε, επιχειρήσει αλλά και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Μόνο εκεί θα δημιουργηθούν κάποιοι θύλακε αριστεία ε, με ανάμειξη διαφόρων φορέων ε, και διαφορεμένων παραγόντων. Με στόχο φυσικά την θέση στην αγορά. Είναι κινητήριο μοχλό η ανάμειξη των ε, τοπικών παραγόντων και θα πρέπει να αναμειχθούν ε, πλήρω στην εφαρμογή του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερε ευθύνε στι τοπικέ και περιφερειακές αρχέ, εξασφαλίζοντα ε, και μακροπρόθεσμα την αρχή τη χρηματοδότηση. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στηρίζεται στην εταιρική σχέση θα πρέπει να εξασφαλιστεί όμως και η χρηματοοικονομική φερεγγιότητα των διαφόρων εταίρων. Και μάλιστα ε, με τις περικοπές που θα γίνουν στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα πρέπει να επιμείνουμε στην ε, χρηστή διακυβέρνηση στα πλαίσια και της κρίσης που μας περιορίζει. Θα πρέπει επίση να διευκρινίσουμε του στόχου του 7ου ερευνητικού προγράμματο πλαισίου. Και τα κονδύλια που θα επενδυθούν θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δεν μπορούμε να διασπαθίζουμε τα δημόσια κονδύλια σε προγράμματα που δεν καταφέρουν να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα. Θα επιμείνω λοιπόν στην έκθεσή μου στην ανάγκη συγκέντρωση τη χρηματοδότηση του 7ου Ερευνητικού Προγράμματο Πλαισίου σε κάποια σχέδια αριστεία και ε, μεγάλη εμβέλεια. Έτσι θα ενισχύσουμε την αξιοπιστία των ε, διαφόρων κοινοτικών μηχανισμών για την ε, πρόθεση της έρευνας. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο θετικό αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών σε ολόκληρη την κοινοτική επικράτεια άσχετα με το επίπεδο επιστημονικής ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών. Προγράμματα αριστείας δεν σημαίνει ότι θα παραμεριστούν όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Η γνωμοδότηση που θα υποβάλω στην Επιτροπή ΙΤΡΕ θα συνδέσει πιο στενά την πολιτική κοινοτομία με την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξη, κάτι που προποθέτει μια αναζήτηση συνεργειών και αποτελεσματικότητας και καλύτερη διακυβέρνηση των ερευνητικών προγραμμάτων μέσω μιας ε, αποκέντρωσης ε, της εφαρμογής του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Αυτά προς το παρόν, ω προς το περιεχόμενο που θα έχει γνωμοδότησή μου. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα σχόλιά σας και τις παρεμβάσεις σας για τη γνωμοδότηση. Ο κύριος Βαν Νίστελ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ με τα λεγόμενα του κυρίου Κεντέκ. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος ε, των ε, ευθυνών μας να δούμε την ε, ε, εδαφική διάσταση σε όλα αυτά τα θέματα. Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω. Όταν ε, σκέφτεται κανείς τα κονδύλια που αφιερώνονται στην έρευνα και στα, στις υποδομές για την έρευνα, καταλαβαίνω ότι πρόκειται για ένα ποσό γύρω στα 50 δισεκατομμύρια για τις ερευνητικές υποδομές, για τα ε, κάμπους τεχνολογίας και αν προσθέσω και τα κονδύλια για την καινοτομία, φτάνουμε στα 85 δισεκατομμύρια. Αν σκεφτούμε τα ποσά που αναφέρονται στο πρόγραμμα πλαίσιο, θα πρέπει να σκεφτούμε Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο μέσα ώστε να έχουμε μια ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ε, στα πλαίσια της έκθεσης για τις συνέργειες ε, έχω κάποιες προτάσεις να κάνω. Θα πρέπει όμως να βασιστούμε στην πρακτική εμπειρία. Κατά την περίοδο αυτή, 2007-2013, σχετικά με το θέμα της συμμετοχής των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, ιδιαίτερα, βλέπουμε μια μεγάλη οπισθοχώρηση. τα πράγματα ήταν το, είναι τόσο πολύπλοκα που οι διαδικασίες είναι τόσο πολύπλοκες που λίγες επιχειρήσεις ε, είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν σε αυτόν τον κυκαιώνα το γραφειοκρατικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε ε, ότι χρειάζεται ε, μία προσέγγιση ε, one stop, ενιαία θηρίδας. Να μην είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να το λύσουμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ και 30 χρόνια μιλάμε για το θέμα του ανοίγματο στην καινοτομία. Ε, οι επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια μπορούν να συμμετέχουν στα μεγάλα προγράμματα, αλλά ε, πάντοτε σε επίπεδο μικρών ε, πρωτοβουλειών Επίση, πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της έρευνα, τη βασική έρευνα, τη εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά θα πρέπει σε όλα αυτά τα νέα προϊόντα, τις νέες διαδικασίες, να λαμβάνεται υπόψη η ε, ε, χωρική διάσταση, η εδαφική διάσταση. Επέμεινα Ε, μάλλον ε, ε, η κυρία Καρβάλιο ακολουθεί μια πολύ ολοκληρωμένη προσέγγιση και νομίζω ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς όμως έχουμε το καθήκον να ενσωματώσουμε την εδαφική διάσταση ώστε να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια, παρατηρήσεις. Αν όχι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με τον προηγούμενο μιλητή. Σωστό είναι η συγχρηματοδότηση να παραμείνει κανόνας. Ε, Βεβαίως τα μεγάλα προγράμματα ε, είναι καλά, αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε αυτά. Αυτό με ανησυχεί αν θέλουμε να περιοριστούμε σε αυτά. Στην ε, κεντρική Ευρώπη και τη χώρα μου την Αυστρία υπάρχουν πολλές μικρές ε, επιχειρήσεις. Η Μεχατρόνικ για παράδειγμα στο Λίντσε δεν είναι μεγάλης κλίμακας ε, βιομηχανικό πρόγραμμα, ούτε έχει μεγάλη βιομηχανική υποστήριξη. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, ε, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούμε στην μεγάλη καινοτόμο δύναμη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα, τις διαδικασίες φιλικότερες προς το χρήστη. Δεν είναι δυνατόν η απόδοση να είναι άριστη αλλά λόγω της γραφειοκρατίας να υπάρχει αποθάρρυνση και να μην ε, παίρνουν την υποστήριξη που δικαιούνται οι επιχειρήσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Αν όχι, παρακαλώ τον εισηγητή να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καθησυχάσω κάπως τον αυστριακό συνάδελφο. Διευκρίνησα ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για πρόθεση των ε, προγραμμάτων αριστείας, αλλά διευκρίνησα επίσης ότι ε, όποιο και αν είναι το επίπεδο επιστημονικής ανάπτυξης, αυτά ισχύουν, άρα δεν εξαιρούμε τα άλλα προγράμματα. Καλό είναι να εστιάσουμε βέβαια στα προγράμματα αριστείας. Όσον αφορά τώρα την εδαφική διάσταση και την περιφερειοποίηση, είναι ένα σημαντικός παράγοντας. Επίσης η εταιρική σχέση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, οι εταιρικέ σχέσεις και κάτι άλλο ε, που δεν τονίστηκε πολύ, ότι ε, θα πρέπει η προσέγγιση να βασίζεται στα αποτελέσματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Το σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη είναι τα διάφορα. Ο κύριος Βαν Νίστελρόι. Με ενδιαφέρει το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε. Στο Βέλγιο είμαστε. Να μας δοθεί το πρόγραμμα της Βελγικής Προεδρίας για την πολιτική συνοχή, ε, ε, έρευνα κλπ. Α, έχω ακούσει ότι υπάρχει. Εμείς μετά θα ενημερώσουμε. Μια μικρή αλλαγή πριν τελειώσουμε που αφορά το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Θυμάστε ότι είπα ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 28 Ιουνίου. Αλλά Χρειάζεται πιο πολύς χρόνος. Και έτσι η προθεσμία δεν είναι 28, είναι η 29η Ιουνίου. 29 Ιουνίου. Συμφωνείτε όλοι. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Uh, Θέλετε κάτι να μας πείτε. Ορίστε. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα εκ μέρους της Ισπανικής Προεδρίας να σας αποχαιρετήσω και να ευχαριστήσω την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για την στενή συνεργασία που είχαμε στο εξάμενο της Ισπανικής Προεδρίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία και η επαφή με την Πρόεδρο και με τα μέλη και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ήταν πολύ αγαστή η συνεργασία και μας ε, βοηθήσατε πραγματικά σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας αποχαιρετήσω εκ μέρους της Ισπανικής Προεδρίας. Ευελπιστώ ότι η αγαστή αυτή συνεργασία θα συνεχιστεί. Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής μας να σας ευχαριστήσω.